just cancelled. So, Mr. Okay. Kérem a kollégákat, hogy aki el szeretne menni a Συνάδελφοι, όσοι θέλουν να φύγουν, παρακαλώ να βγουν από την αίθουσα γρήγορα και ήσυχα κυρίως για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με τις αιτιολογήσεις ε, ψήφου. Συνάδελφοι, η πρώτη έκθεση είναι επιμελητεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Πολυτροπικέ Μεταφορέ. Ο κ. Πόσπισιλ έχει τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και θα προσπαθήσω να εξηγήσω γιατί ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής. Πιστεύω λοιπόν ότι η έκθεση αυτή θα